ευχαριστώ που με βοηθάτε να πολεμήσω σε αυτή τη μάχη που δίνω. Ευχαριστώ. Ε, με αυτήν ε, την τελική θέση κλείνει η συζήτηση. Αύριο στις 12 η ώρα έχουμε την ψηφοφορία. Περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα της μερίσιας διάταξης, ε, την έκθεση Μιλντερ για την κυκλοφορία στην αγορά και χρήση πρόδρομων ουσιών ουσιών εκρηκτικών υλών. Ζητώ λοιπόν, ε, δίνω λοιπόν το λόγο στον κύριο Μούλτερ. De commissie, het voorstel van de commissie over dit onderwerp kwam reeds. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ταιριάζει Μάλλον ήρθε την εποχή που διαμορφώθηκαν εκείνα, υπήρξαν και τα γεγονότα στην Νορβηγία. Είναι σημαντικό να υπάρχουν κανόνες σε αυτόν τον τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε ύλε που μπορούν να ε, χρησιμοποιηθούν για κατασκευή εκρηκτικών θα πρέπει να ρυθμίζονται για να αποφεύγονται προβλήματα στο μέλλον. Γι' αυτό πρότεινε κανονισμό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι οδηγία. Ούτως ώστε να έχουμε κοινούς κανόνες και να συμμορφώνται τα κράτη-μέλη με αυτούς τους κανόνες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο συμφωνούν. Το Συμβούλιο όμως φαίνεται να διαφωνεί. Κάποιες χώρες έχουν σύστημα καταχώρησης και όχι αδειοδότησης. Σαν Κοινοβούλιο είμαστε ικανοποιημένοι με τον συμβιβασμό αυτό στον οποίο καταλήξαμε μετά από πέντε χρόνια να γίνει αναθεώρηση ούτω ώστε να δούμε πώς λειτουργούν τα διάφορα συστήματα και στο τέλος να έχουμε ένα ενίο σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποφασίστηκε ένας προκατακτικός κατάλογος, αρχικός κατάλογος περιορισμένου αριθμού ουσιών σε συγκεντρωμένες συγκεντρώσεις που μπορούν να αγοραστούν με άδεια και μόνο ένας κατάλογος αυτός. Και έχουμε άλλο κατάλογο ε, για ουσίες για τις οποίες αν υπάρχουν κάποιες υπόνοιες θα πρέπει να εξεταστούν. Θα πρέπει να υπάρχουν και σημεία επαφής στις χώρες ούτως ώστε να καταχωρούνται διάφορες συναλλαγές και αγοροπολισίες των ουσιών αυτών και να μπορούν να αντιδρούν το ταχύτερο δυνατόν τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω λοιπόν ότι το, η θέση του Κοινοβουλίου όσον αφορά τον καθορισμό των υπόπτων συναλλαγών ε, είναι μια βελτιωμένη προσέγγιση θα πρέπει συνεχώς να υπαγρυπνούμε όσον αφορά τις ουσίες και στον κανονισμό συμπεριλαμβάνεται και η ιδέα ε, μιας διαβούλευσης με τα κράτη-μέλη και τους εμπειρογνώμονες σχετικά με το θέμα. Αν χρειάζεται τροποποίηση του καταλόγου, να μπορεί να, να γίνεται αναθεώρηση. Έκανε μια τέτοια παραχώρηση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εάν μπορούν να αποσυρθούν ή να μπουν νέες στον κατάλογο. Αυτό για να γίνει πρέπει να γίνει μέσω διαδικασίας νομοθετικής η προσθήκη αφαίρεση ουσιών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτιμούσε κατά εξουσιοδότηση πράξη, αλλά δεν μπορούμε να πετύχουμε όλα όσα θέλουμε. Το Συμβούλιο ε, τελικά επεκράτησε όσον αφορά τη θέση του για το συγκεκριμένο θέμα. Όσον αφορά τις συγκεντρώσεις, οι κατεξουδότηση πράξεις εφαρμόζονται και μπορεί το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να συμφωνήσουν ή να μην συμφωνήσουν. Όσον αφορά το ζωτούχο αμμόνιο, συμφωνούμε. Καλύπτεται το πεδίο εφαρμογής του REACH. Μακροπρόθεσμα συμφωνούμε να γίνει μια αξιολόγηση. Μήπως θα έπρεπε να ενταχθεί και αυτή η ουσία στα πλαίσια του παρόντος κανονισμού. Όσον αφορά τους ελέγχους, οι έλεγχοι θα, διεξάγονται από τα, θα διενεργούνται από τα κράτη-μέλη. Θα επιβάλλονται πρόστιμα σε περιπτώσεις παραβάσεων που θα προβλέπονται κυρώσεις από τα κράτη-μέλη και θα πρέπει ε, τα, οι κυρώσεις οικονομικές, τα πρόστιμα να είναι επαρκή. Νομίζω ότι κάνουμε ένα βήμα προς σωστή κατεύθυνση για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την πρόληψη μείωση του κινδύνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε τον εισηγητή για την Κομισιόν, η κυρία Ρέντινγκ. Πρόεδρε, πιστεύω ότι όλοι γνωρίζουμε ποιος είναι ο ε, κίνδυνος ασφαλείας ε, που ε, συνιστούν οι τρομοκράτες. Δεν χρειάζεται να σας υπενθυμίσω τα τελευταία χρόνια πόσες ζωές έχουν χαθεί άδικα και άκρητα λόγω τρομοκρατικών ενεργείων. Θα πρέπει από διάφορες πλευρές να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα. Σήμερα πραγματευόμαστε μία μονοδιάσταση. Πώς να δυσκολεύσουμε τη ζωή των βίων εξτρεμιστών ως προς την πρόσβαση που έχουν σε πρόδρομες ουσίες για την κατασκευή ε, εκρηκτικών υλών. Ο στόχος ήταν να εναρμονίσουμε τους κανόνες, να μειώσουμε την πρόσβαση του κοινού σε πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών ε, και να μην μπορούν έτσι να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή παράνομων εκρηκτικών. Ε, καθίσταται λοιπόν ε, έκνομη παραγωγή, η αγορά και αυτών των πρόδρομων ουσιών και παραγωγή εκρηκτικών υλών. Προστατεύουμε, ε, συγγνώμη, επιρρύπουμε το, την ευθύνη και το βάρος στους πολιτές και στους παραγωγούς και τους μεταπολιτές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους μετέχοντες, τα τρία θεσμικά όργανα για τις προσπάθειες που έχουν κάνει. Πρόκειται για συμφωνία των νομοθετών ναι, και το εγκεκριμένο σχέδιο θα βελτιώσει σημαντικά την ασφάλεια στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και θα προσφέρει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Ε, ε, εξακολουθεί να υπάρχει όμως ένα μήλο της έρηδος η πράξη σε και θα ήθελα επ' αυτού να κάνω μια δήλωση από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή σημειώνει τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι συνομοθέτες για το άρθρο 9.1 καθώς και την ομοφωνία ε, που επήλθε στο Συμβούλιο. Υπενθυμίζει όμως ότι το άρθρο 290 πρέπει να ερμηνευτεί ως εξής. Ε, διαθέτει αυτονομία Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, προετοιμασία και κατάρτιση πράξεων κατεξουσιοδότηση. Η συμφωνία των τριών θεσμικών οργάνων απηχεί αυτήν την αρχή και περαιτέρω θα πρέπει σε μια αιτιολογική σκέψη και όχι στο διατακτικό να αναφέρεται οποιαδήποτε γνωμοδότηση εμπρογνωμόνων. Λυπούμεθα που δεν τηρήθηκε αυτή η αρχή και τονίζουμε ότι η τωρινή υπόθεση σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελέσει νομικό προηγούμενο. Ελπίζουμε πάντως ε, ότι αύριο θα είναι θετική η έκβαση της ψηφοφορίας, ώστε το Συμβούλιο επισήμως να μπορέσει να εγκρίνει το νέο νομοθέτημα πριν από το πέρας ε, του τρέχοντος έτους ε, και θα κάνουμε και εμείς αυτό που μας αναλογεί, δηλαδή θα εκδώσουμε κατευθυντήριες γραμμές σε σχέση με την εφαρμογή πρώτου να αρχίσουν να ισχύουν οι κανόνες, δηλαδή 18 μήνες μετά τη θέση ισχύ του κανονισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την Επίτροπο. Έχει ζητήσει τον ε, λόγο η κυρία Αναμαρία Κοράτσα Μπίλτ. Το καλοκαίρι το ελληνικό του 2011 συγκλονιστήκαμε όλοι. Γιατί μάθαμε ότι στην Ορβηγία, σε ένα νησί, όπου είχα μαζευτεί νέοι, διεπράγει μια σφαγή στην καρδιά του Όσλο. Και η καρδιά του Όσλο ήταν ε, θύμα βομβιστικής επίθεσης. Σύμφωνα με την Ευρωπόλ, ένας από τους βασικούς λόγους για τον οποίο ε, βρήκαμε τον ένοχο είναι διότι αγόραζε πολλές χημικές ουσίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ε, ετοιμασία εκρηκτικών υλών, κατασκευή εκρηκτικών στο σπίτι. Είναι ευπρόσδεκτο που τελικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα κράτη-μέλη και ελπίζω και το σώμα να συμφωνήσει ε, και έχουμε καταλήξει σε μια πολύ καλή πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναρμόνιση των κανόνων που υπάρχουν τώρα για την πρόληψη τέτοιων ε, φρικτών γεγονότων. Δεν θέλουμε να επαναληφθούν αυτό και αυτά. Η τρομοκρατία, η εγκληματικότητα είναι διασυνοριακή. Οι κανόνες μας είναι διαφορετικοί και κατακαιρματισμένοι. Τι μπορούμε να κάνουμε για να προχωρήσουμε. Πρώτα απ' όλα στα περισσοτερα κάτι κράτη-μέλη θα υπάρχει ανάγκη άδεια για να μπορεί κάποιο να αγοράσει από ένα χονδρέμπορο, από κάποιο κατάστημα, αυτά τα εκρηκτικά, αυτέ τι ουσίε, τι πρόδρομε ουσίε. Αυτέ τι χημικέ ουσίε, οι οποίε μέχρι κάποια συγκέντρωση, κάποιο κατόφλι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, γιατί σε αυτέ τι συγκεντρώσει που να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή εκρηκτικών. Μετά, με την νομοθεσία αυτή εξασφαλίζουμε ανιχνευσιμότητα. Οπότε οι εμπορευόμενοι θα πρέπει να ενημερώνουν όταν πολλούν ε, μεγάλες ποσότητες αυτών των ουσιών. Και έχουμε καλό σύστημα προστασίας των δεδομένων όσον αφορά τις συναλλαγές αυτές που πρέπει να αναφέρονται. Και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να καθορίσουν τις κυρώσεις που θα επιβάλλουν σε περιπτώσεις παραβάσεων. Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα κύριε Πρόεδρε, και σε τρία χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μα πει: Χρειάζεται να προχωρήσουμε πιο πέρα, χρειάζεται περαιτέρω εναρμόνιση. Και καλό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυ κατά πόσο οι κανόνε που εγκρίνουμε τώρα είναι επαρκεί, αν αρκούν, ούτω ώστε να εξασφαλίζουν την ασφάλεια των πολιτών μα. Έχουμε πετύχει, πιστεύω, τη σωστή ισορροπία. Έχουμε ασφάλεια από τη μία πλευρά, που ήταν πρωταρχική μα μέρημνα, και απ' την άλλη μη αύξηση της γραφειοκρατίας για τους αγρότες, για τις εταιρείε, για τα ξενοδοχεία που έχουν πισίνες που χρειάζονται χημικά για να καθαριστούν και έχουμε ισορροπία μεταξύ υποβολής αναφορών, ενημέρωσης και προστασία των δεδομένων. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα πραγματικά να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω τον τη σκιώδη συγγήτρια, την κυρία Βερονίκ του ΕΛΚ, που δυστυχώς ταυτόχρονα ως συντονίστρια πρέπει να είναι σε πολύ, μια πολύ σημαντική άλλη συνάντηση η εγκληματικότητα. Αλλά απίλευσε τη συνεργασία με τον συγητή. Πιστεύουμε ότι έκανε το κάτι παραπάνω. Αυτό πιστεύουμε στο ΕΛΚ. Έδειξε ευελιξία και συμφώνησε με τους άλλους γιατί είναι σημαντικότατο το νομοθέτημα αυτό για την αποφυγή της τρομοκρατίας και της εγκληματικότητας και προστατεύει και τους πολίτες στην Ευρώπη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κυρία Γκόμες τώρα. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για τον προσανατολισμό που ακολούθησε, την προσήλωση, την αφοσίωσή του και την αγαστή συνεργασία με όλους τους κυριώδες εισηγητές. Αυτό η νέα πρόταση προστατεύει τους πολίτες διότι περιορίζει την πρόσβαση και ελέγχει τις συναλλαγές με τις επικίνδυνες πρόδομες ουσίες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή εκρηκτικών υλών. Έχουμε πολλά παραδείγματα τέτοιων οικιακών βομβών στην Ευρώπη και δεν καταλαβαίνω γιατί το Συμβουλίο, γιατί τα κράτη-μέλη χρειάστηκαν τόσο χρόνο για να καταλήξουν σε, μια, σε ένα συμβιβασμό με το Κοινοβούλιο ούτω ώστε να μπορέσουμε να εγκρίνουμε επιτέλους την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, η επίθεση Μπρεβίκ στην Νορβηγία έγινε όντω με ένα τέτοιο αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό και ε, κατέστη απαραίτητο να πάρουμε στα σοβαρά την ασφάλεια των πολιτών ε, και να ρυθμίσουμε και τις αναλλαγές ε, φυσικών και νομικών προσώπων. Ε, τώρα, τα συστήματα διοδότησης με διαφέρουν από κράτο σε κράτος και η Νορβηγία ισχυρίζεται ότι το σύστημα καταχώρησης και το σύστημα διοδότησης που έχει λειτουργεί αισίως. Η προτεραιότητα θα πρέπει να αποδοθεί στην προστασία των πολιτών διότι δίνουμε τροφή στους τρομοκράτες ε, ε, θα πρέπει ταχύτατα να εγκριθεί αυτό το νομοθέτημα, να μεταγραφεί το νομοθέτημα στην εθνική νομοθεσία, ούτω ώστε ε, τα νέα εθνικά συστήματα να υπάγονται στις νέες ευρωπαϊκές σε γραμμές για τις πρόδρομες ε, ουσίες των εκρηκτικών υλών. Καλύπτονται 8 ουσίες μέσα στον κανονισμό, αλλά το θέμα εδώ δεν είναι η εμπορευματοποίηση, η αγορά ή η αδειοδότηση των εκρηκτικών ουσιών. Θέλουμε να να αυξήσουμε την ασφάλεια ως προς την πρόσβαση και την χρήση ε, ειδικών ουσιών γενικής χρήσης ε, που χρησιμοποιούνται όμως για επικίνδυνους σκοπούς. Ε, θέλουμε μεγαλύτερη χνηλασιμότητα για να αποφύγουμε τις τραγωδίες της Νορβηγίας το 2011 ή του Λονδίνου το 2005. Σας ευχαριστούμε κύριος Άλμπρεχτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, να ευχαριστήσω εξηγητή για την πολύ καλή εργασία του. Είναι ξεκάθαρο ε, που πρέπει να ε, επέβουμε όταν μιλάμε για τον αγώνα κατά της τροποκρατίας. Στην καθημερινή ζωή είναι σημαντικό να δίνουμε στους ανθρώπους να καταλάβουν που βρίσκεται ο κίνδυνος για τέτοιες ε, επιθέσεις, για εγκληματικότητα, έτσι ώστε ε, να είμαστε ασφαλείς όταν μιλάμε για όπλα αλλά και για εκρηκτικές ουσίες σαν αυτές για τις οποίες μιλάμε σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μπορούμε να πούμε ότι ε, δεν μπορεί κανείς να έχει ανα πάσα στιγμή άμεση πρόσβαση χωρίς περιορισμούς σε εκρηκτικές ουσίες ή σε ουσίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ε, δημιουργία εκρηκτικών υλών. Ε, θα πρέπει να υπάρχει κάποια καταγραφή ε, δεν είναι και μεγάλο πρόβλημα να καταγράφεται ποιος αγοράζει αυτές τις ουσίες έτσι ώστε να μπορεί να δικαιολογήσει γιατί τις χρειάζεται ας πούμε, για την περαιτέρω επεξεργασία αυτών για συγκεκριμένους δηλωμένου σκοπού. Υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένε ομάδε, όπως είπε και η κυρία Κορέτσα Μπίλτ, που ε, δεν πρέπει να εμποδίζονται να αγοράζουν μικρές ποσότητε αυτών των ουσιών για άλλους σκοπού. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να προσέξουμε ε, να υπάρχει ένα σύστημα ασφαλείας που θα λαμβάνει ε, υπόψη όλες αυτές τις περιπτώσεις έτσι ε, ώστε να ε, γίνεται και συλλογή στοιχείων που είναι σημαντική για να μπορέσουμε να προειδοποιούμε για περιπτώσεις που μπορεί να είναι επικίνδυνες. Ευχαριστώ λοιπόν για τη συμβολή όλων, αλλά και να επαναλάβω αυτό που είπα, είναι πολύ σημαντικό να επιστήσουμε την προσοχή για τον κίνδυνο ειδικότερα ε, ώστε να, για τέτοια θέματα ε, τα οποία θα μας βοηθήσουν να μειώσουμε τις δυνατότητες που δίνονται σε ανθρώπους που θέλουν να κάνουν τρομοκρατικές ενέργειες, να κάνουν τέτοιες ενέργειες και να μπορούμε να αντιδρούμε ε, σωστά και όχι με μέτρα ε, παρακολούθησης. Αυτό είναι το σημαντικό και γι' αυτό υποστηρίζω αυτό το μέτρο, οι πράσινοι υποστηρίζουν αυτό το μέτρο και χαιρόμαστε που μπόρεσε να έρθει ε, σε αυτή την ε, Επιτροπή. Ευχαριστούμε η κυρία Φλαζικόφα Μπένοφα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, η Επιτροπή έχει θεσπίσει ένα σχέδιο δράσης ε, για την διασφάλιση των εκρηκτικών υλών. Έχουμε την Επιτροπή, η οποία αποφάσισε για τις πρόδρομες ουσίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε τρομοκρατικές επιθέσεις. Κάποια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έχουν ε, ήδη θεσπίσει νόμους σχετικά με τις ουσίες που μπορούν να μπουν στην, που υπάρχουν στην αγορά οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως πρόδρομες ουσίες για εκρηκτικά. Είναι πολύ σημαντικό ε, λοιπόν να υπάρχει συγκεκριμένη ρύθμιση αυτών και να εναρμονιστούν και οι κανόνες έτσι ώστε η ελεύθερη ε, το ελεύθερο εμπόριο να ε, απλουστευτεί, αλλά ε, και η πρόταση της Κομισιόν θα πρέπει να εμποδίζει ε, στο ευρύ κοινό να έχει πρόσβαση σε τέτοιες ουσίες που μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως πρόδρομες ουσίες για εκρηκτικά. Θα πρέπει έτσι με αυτόν τον τρόπο να μειώσουμε και τη συχνότητα αλλά και το μέγεθος των τρομοκρατικών επιθέσεων. Είναι σημαντικό ε, ταυτόχρονα βέβαια να διασφαλίσουμε και την προσωπική σφαίρα του καθενός, τα προσωπικά δικαιώματα, έτσι ώστε ε, ε, και, και να μπορούμε να αντιδρούμε εγκαίρως όταν χρειάζεται. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε λάβει υπόψη μας και τη θέση του πολίτη. Γι' αυτό υποστηρίζω την, ε, τον κανονισμό για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ερχόμαστε στη διαδικασία Catch the Eye. Έχουμε δύο αιτήματα για αυθόρμητες ε, παρεμβάσεις. Κυρία Μπασέσκο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είναι σημαντικότατος αυστηρός έλεγχος των προδρόμων ουσιών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή αυτοσχεδίων βομβών, για την προστασία και της ενώσεως και των πολιτών της. Ξέρετε, αυτά τα εκρηκτικά είναι το αγαπημένο εργαλείο των τρομοκρατών. Πέρσι, στην βομβιστική απόπειρα, βομβιστική επίθεση που έγινε στο Όσλο, χρησιμοποιήθηκαν ουσίε όπω ε, το άζωτο τη ε, μονιούχο άζωτο, που συμπεριλαμβάνεται στο παράρτημα τη προτάσεω κανονισμού για να αποφευθεί η επανάληψη τέτοιων τραγωδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να κινηθούμε προσεκτικά. Αυτές οι ουσίες δεν θα πρέπει να διατίθενται στο εμπόριο χωρίς άδεια και τέτοιες πρακτικές θα πρέπει να αποθαρρύνονται από τα κράτη-μέλη. Οι εθνικές αρχές θα πρέπει συνεχώς να ελέγχουν τις άδειες που χορηγούνται. Επίσης και θελοντική επισήμανση των, υπο... των ε, συναλλαγών θα είναι κάτι που θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο για να αποφευχθούν επικίνδυνες καταστάσεις. Ευχαριστώ κύριε uh, Ευχαριστώ. Ασύνηθε παράδειγμα αυτό είναι ότι αναγνωρίζει ένα πραγματικό πρόβλημα η Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί διεθνώ αλλά όχι απαραίτητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόβλημα ψηφίσεω νόμου που απαγορεύει τον κόσμο τον μπορεί να αγοράζει κάτι είναι ότι όσο πιο περισσότερο χρόνο χρειάζεται η διαδικασία, τόσο μεγαλύτερε πιθανότητε ο αγοραστή και σε αυτή, την σε αυτή την περίπτωση ο τρομοκράτη να μαζεύει σιγά σιγά, να συσσωρεύει από πριν, πριν γίνει η απαγόρευση τη ουσία. Το θυμάμαι εδώ στην Επιτροπή Λίμπε πριν από ένα χρόνο είχε αναφερθεί και δεν ξέρουμε και πότε θα περάσει τελικά η νομοθεσία και πότε θα τεθεί σε ισχύ. Θα ήταν προτιμότερο να είχαμε συμφωνήσει σε διεθνέ επίπεδο, να ζητήσουμε την υποστήριξη βιομηχανία και να υπάρχει ένα εθελοντικό δελοντουργικό κώδικα που θα εφαρμόζεται και θα ρίχνουμε τα όλε τι χώρε συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών να θεσπίσουν νομοθεσία αμέσω. Το Ηνωμένο Βασίλειο, στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί κανεί σε κάποιε περιπτώσει να ψηφίζει νομοσχέδιο εντό 24 ώρου. Η διαδικασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι μακρά και λεπτομερής και είναι απίθανο κάποιοι που να μην έχουν μαζέψει όλες, να μην έχουν συσσωρεύσει αυτές τις ουσίες οι, αυτοί που θέλουν να διαπράξουν κάτι τέτοιο εκ των προτέρων πριν θεσπιστεί η νομοθεσία. Um, ε, αυτή η έκθεση σχετίζεται με τον κανονισμό που έχει ως στόχο την παρεμπόδιση της ε, πρόσβασης, εύκολης πρόσβασης σε ένα μεγάλο αριθμό ουσιών ε, που χρησιμοποιούνται για σύνομους σκοπούς σε μεγάλο βαθμό. Δυστυχώς στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε εκτεταμένη εμπειρία στους αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς. Παραδείγματος χάρη χρησιμοποιεί τη βάση λοιπασμάτων από τους τρομοκράτες εδώ και χρόνια για την κατασκευή τέτοιων μηχανισμών ε, και πρόκειται για έναν κανονισμό που στόχο έχει να διευρύνει την αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιώντας ως πρόφαση ε, την αποτροπή των τρομοκρατικών ενεργειών. Γι' αυτό οι συναδελφοί μου και εγώ θα καταψηφίσουμε αυτό το, αυτή την πρόταση. Σας ευχαριστούμε. Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομη, Πρόεδρε διότι όλοι οι λογικοί άνθρωποι εδώ στο Κοινοβούλιο συνειδητοποιούν ότι χάρη σε αυτόν τον κανονισμό θα κάνουμε ένα σημαντικό βήμα και θα υποδείσουμε τους τρομοκράτες ώστε να μην προμηθεύονται εύκολα τις ουσίες για την παραγωγή αυτοσχεδίων εκρηκτικών μηχανισμών. Θα προστατεύσουμε έτσι τις χώρες μας και με αυτόν τον κανονισμό όντω αναβαθμίζεται η δημόσια ασφάλεια και απλουστεύεται το ζήτημα και για τους προμήθευτές διότι θεσπίζεται ένα εναρμονισμένο σετ κανόνων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει η Ένωση της εργασίας και σε άλλους τομείς για την μείωση των απειλών της τρομοκρατίας. Θα σα δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, παραδείγματο χάρη ε, το δίκτυο για τη συνειδητοποίηση της ριζο παστικοποίηση ε, που επιτρέπει ανταλλαγή εμπειριών επιτόπου για ανθρώπους που ενδέχεται να ε, μεταπιστούν, να εμπλακούν σε τέτοιες ε, τρομοκρατικές ε, ενέργειες. Έδωσα αυτό το παράδειγμα για να σας δείξω ότι αντιμετωπίζουμε αυτό το θέμα από διάφορες πλευρές. Κύριε Μούλτερ επιτρέπεται κάποιος που ήρθε αργά και δεν ήταν στον κατάλογο των ομιλητών ε, να μιλήσει και μετά να μιλήσετε εσείς. Ευχαριστώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ που με παρατηρήσατε, που με είδατε, παρόλο που άργησα να σηκώσω το χέρι μου. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και νομίζω ότι θα πρέπει να συζητήσουμε αυτόν τον κίνδυνο που ελοχεύει όλο και περισσότεροι εξτρεμιστές έχουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους. Όμως, κυρία Επίτροπε, πιστεύω ότι θα ήταν σόφρον να επεκτείνουμε αυτή την προσέγγιση και σε άλλους τομείς που δεν συνδέονται με την τρομοκρατία αυτή καθεαυτή αλλά με την ασφάλεια ή με διάφορες τάσεις για βία. Παραδείγματος χάρη ε, τα όπλα ε, μπορεί κάποιος να αγοράσει όπλο και είναι σαφές ότι η εγκληματικότητα αυξάνεται στον κόσμο και είναι ξεκάθαρο για μένα ότι αυτό ε, σχετίζεται με την κατοχή όπλων και την εύκολη πρόσβαση στα όπλα. Πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον ε, εισηγητής παρακαλώ το λόγο. Ευχαριστώ όλους εκείνους που συμμετείχαν σε αυτή τη συζήτηση και θα ήθελα να χρησιμοποιήσω αυτή την ευκαιρία να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης εισηγητές για την συνεργασία τους. Ήτανε... Έχω υπέροχες αναμνήσεις από τη συνεργασία. Ε, πιστεύω ότι όλοι έκαναν κάθε προσπάθεια και κατάφεραν στο τελικό αποτέλεσμα να αντικατοπτρίζονται οι απόψει του. Ε, ξέρω ή γνώριζα μάλλον ότι ήταν δύσκολο σημείο αυτό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χρειάστηκαν όμως τελικά παραχωρήσεις από όλους για να καταλήξουμε σε κάποιο αποτέλεσμα. Ε, λοιπόν, λέει ότι εδώ θα πρέπει να γίνεται προσπάθεια για διαβούλευση με τους εμπειρογνώμονες. Endeavor στα αγγλικά, προσπάθεια λέει ότι θα γίνεται στο μέλλον για διαβούλευση με τους εμπειρογνώμονες. Αυτό είναι κάτι που επελέγει για να αφήσουμε μεγαλύτερο περιθώριο επιλογής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν θα ψηφίσουμε αύριο ε, το κείμενο αυτό, δεν μπορώ να εγγυηθώ 100% ότι θα επιτύχουμε μετά την ψηφοφορία 100% ασφάλεια για τους πολίτες όσον αφορά αυτές τις ουσίες. Πιστεύουμε όμως ότι κάναμε σωστό βήμα με αυτή την πρόταση για να αποφύγουμε και άλλες απόπειρες τρομοκρατικές ενέργειες. Ευχαριστούμε τον εισηγητή. Κλείνει η συζήτηση για αυτό το θέμα. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 12. Ερχόμαστε τώρα στις ε,